Έλαβα από την ομάδα των φιλολευθέρων ορισμούς ε, για τα μέλη μιας επιτροπής και μιας αντιπροσωπείας. Ε, αυτά θα αναφέρονται στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης και αν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση από την ε,